του κυρίου Γεώργιου Κίρτσου και του κυρίου Στέλιου Κούλογλου σε ό,τι αφορά δύο ποινικέ διαδικασίε, οι αρμόδιε αρχέ ζήτησαν επίση ε, την άρση τη ε, ασυλία του κυρίου Ρόμπερτ Ιβασκεύσκη και του κυρίου Σικέρσκη. Και σύμφωνα με τον κανονισμό, αυτά παραπέμφθηκαν στι αρμόδιε ε, νομικέ στην Επιτροπή